είναι διαδικαστικό. Κάνατε πριν διαδικαστικό και νομίζω ότι διευκρίνησε τη διαδικασία Catch Περί τίνος πρόκειται. Αν είναι για το Catch δεν θα δεχτώ το διαδικαστικό. Σωστά είπατε ότι είναι προνόμιο του Προεδρού. Οπότε, ποια θα είναι η δικιά σα πολιτική κατά τη διάρκεια αυτή τη συζήτηση για την μπλε κάρτα. Θα πάρετε δύο, μία ε, και στο Catch ή όχι. Να ξέρω. Νομίζω ότι είναι λογικό που το ρωτάω. Γιατί οι ευρωβουλευτέ, όπω βλέπετε, εκνευρίζονται με την κατάσταση έτσι όπως έχει. Πρόεδρος, κύριε Γκέλ, κατάλαβα την ερώτησή σας. Μόλις έφτασα, όπως είδατε. Δεν έχω δει ακόμα τον κατάλογο. Θα τον κοιτάξω. Θα κοιτάξω και τι ώρα είναι και θα αποφασίσω κατά πόσο θα πάρω μπλε κάρτες ή όχι. Τότε αν θα πάρω μία, δύο ή μόνο για τους εκπροσώπους των ομάδων, ένας σαν ομάδα κλπ. Θα δω. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Επιτρέψτε μου να αρχίσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μου δίνει να έχουμε τη συζήτηση αυτή για την Ανατολική Εταιρική Σχέση ακριβώς πριν από τη διάσκεψη κορυφής της Ρήγα, όπου οι ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης θα συναντηθούν στη Ρήγα 21 και 22 Μαΐου. Έξι χρόνια πριν στην Πράγα μοιραστήκαμε το όρομά μας για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους μας από την Ανατολική Ευρώπη, εμβαθύνοντας περισσότερο στις σχέσεις μας και χτίζοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας και διαλόγου. Έκτοτε, πετύχαμε καλή πρόοδο στην εταιρική μας αυτή σχέση. Υπάρχει καλύτερη κατανόηση των ε, διαφόρων συμφερόντων, των αναγκών και των φιλοδοξιών των εταίρων μας στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Στη Ρίγα λοιπόν θα διαπιστώσουμε τα επιτεύγματα αυτά που έχουμε διαπιστώσει μετά το Βίλνιους και θα καταρτήσουμε μια θετική ατζέντα για το μέλλον. Μετά την ε, προηγούμενη διάσκεψη εταιρική σχέση του Βίλνιους υπογράφτηκε η Συμφωνία Σύνδεσης και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και έτσι φτάσαμε σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας με τη Γεωργία, τη Μολδοβία και την Ουκρανία. Η Συμφωνία Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένη τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τη Γεωργία και τη Μολδοβία, ήδη προσωρινά εφαρμόζονται και τα αρχικά δείγματα είναι πολλά υποσχόμενα. Το εμπόριο έχει αυξηθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους αυτούς. Όσον αφορά την Ουκρανία, η πρόσφατη διάσκεψη κορυφής με την ε, Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε την προσωρινή εφαρμογή της Ουκρανικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με έναρξη την 1η Ιανουαρίου του 2016. Όπως γνωρίζετε, η Επίτροπος Ασίλια Μάλμστρομ έχει τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και την Ρωσία προκειμένου να διασφαλίσει ότι η προσωρινή εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου θα λάβει πράγματι χώρα και κάτω από τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες. Η διάσκεψη της Ρήγας θα λαβει πραγματι χωρα και κατω απο τις καλυτερες δυνατον η διασκεψη της ρηγας θα αποτελεσει μια ευκαιρία για να ξαναδούμε τα πρώτα στάδια της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης και της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εμβαθύνει τη συνεργασία αυτή. Η διάσκεψη θα επιβεβαιώσει τη σημασία που έχουν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες δίνουν μεγαλύτερο βάρος ακόμα στο κράτος δικαίου και στην ανταγωνιστικότητα της, της ε, αγοράς που βασίζεται στην οικονομία και θα διασφαλίσει το ευρωπαϊκό μέλλον των εταίρων μας. Θέλουμε να δείξουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει για μας η οικοδόμηση θεσμών, η κινητικότητα, οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων, οι ευκαιρίες της αγοράς και διασυνδέσεις. Συνεπώς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στο περιθώριο της διάσκεψης αυτής τρεις εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα. Πρώτον, είναι η διάσκεψη για τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Δεύτερον, θα είναι η διάσκεψη για την κοινωνία των πολιτών. Και τρίτον, το Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές θα υπογραμμίσουν τον αυξανόμενο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των ε, επαφών μεταξύ επιχειρήσεων που αποτελούν πολύ βασικό στοιχείο της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι οι ευρωπαϊκές αξίες, οι σχέσεις μας με τις έξι χώρες εταίρους μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας. Για τους εταίρους μας ο δρόμος είναι αυτός. Για ορισμένους είναι άλλες συμφωνίες. Για άλλες χώρες υπάρχει ακόμα περιθώριο δουλειάς. Έχουμε προχωρήσει επίσης σε κατανόηση με την, Αρμανία, με την Αρμενία στα πλαίσια των μελλοντικών μας σχέσεων και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να έχει διαπραγματεύσεις για νέες συμβατικές συμφωνίες με την Αρμενία. Η εντολή ετοιμάζεται τώρα. Όσον αφορά το Αζερμπαϊτζάν, περιμένουμε τις ιδέες του και το πώς βλέπει το μέλλον του και τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν θα έχουμε πάρει τα στοιχεία αυτά, θα δούμε τι είδους σχέσεις είναι καλύτερες και έχουν ανάγκη οι δύο πλευρές. Επίσης, εξετάζουμε πώς θα βαθύνουμε περισσότερο στις σχέσεις μας με τη Λευκορωσία. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ανάπτυξη διμερών σχέσεων με διαφορετικό τρόπο με κάθε χώρα είναι και ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε για τους έξι εταίρους το ενδιαφέρον τους για την ανατολική εταιρική σχέση. Και αυτό ακριβώς το πλαίσιο είναι που επιθυμούμε. Έχουμε προχωρήσει και στο τομέα της κινητικότητας. Από τον Απρίλιο της περσινής χρονιάς η Μολδοβία συμμετέχει σε ένα καθεστώς χωρίς θεωρήσεις στα πλαίσια του Σέγγεν. Κάπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι υποφελήθηκαν. Τώρα και η Γεωργία και η Ουκρανία έχουν προχωρήσει πολύ στην εφαρμογή των κριτηρίων όσον αφορά το καθεστώς ελευθέρωσης θεωρήσεων. Εφόσον ε, τηρούνται οι προϋποθέσεις, στην έκθεση πρόοδου της Επιτροπής οι δύο χώρες αυτές θα μπορέσουν να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Πετροπή εξακολουθεί να ελέγχει και να κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τις χώρες αυτές και θα αναφέρει για την πρόοδό του στα τέλη του 2015. Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων τώρα με τη Λευκορωσία όσον αφορά την Συμφωνία για τη Διευκόλυνση Θεωρήσεων και Επανεσδοχής προβλέπονται επίσης για τον Ιούνιο αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω εδώ ότι η ανατολική εταιρική σχέση και η διάσκεψη αυτή στη Ρήγα λαμβάνει η χώρα μέσα σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου τα σύνορα έχουν αλλάξει δια της βίας και όπου εταίροι και πράγματι χώρες μέλη έχουν υποβληθεί σε σημαντικές πιέσεις. Ε, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω και πάλι ότι δεν συμφωνούμε με την μηδενική βάση κονδυλίων ή για την χρήση της δωροδοκίας. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής. Ούτε η ανατολική εταιρική σχέση, ούτε οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιων εταίρων έχει ποτέ ή στο μέλλον πρόκειται να κατευθυνθεί εναντίον κάποιου αλλά θέλω να είμαι εξίσου σαφής για το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει τους εταίρους μας για να κάνουν ελεύθερες επιλογές όσον αφορά την εξωτερική τους και την εμπορική τους πολιτική. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Και η διάσκεψη στη Ρήγα είναι μια ευκαιρία προκειμένου να ακούσουμε τις απόψεις των εταίρων μας για το μέλλον της ανατολικής εταιρικής αυτής σχέσης. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι επανασχεδιάζοντας την πολιτική μας για το μέλλον έχουμε ακούσει τους εταίρους μας και έχουμε λάβει υπόψη τις δικές τους θέσεις. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, θέλω να επαναλάβω ότι προσφέρουμε στους εταίρους μας της ανατολικής εταιρικής σχέσης μια πραγματική εταιρική σχέση. Δεν επιβάλλουμε επιλογές στους εταίρους μας. Η διαφοροποίηση στις διμερείς μας σχέσεις θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί παρετέρω για να λάβουμε υπόψη μας τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες του καθετέρου. Η πλήρης δέσμευση των κυβερνήσεων των εταίρων μας είναι επίσης ζωτική σημασία για να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Όμως καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πετύχει ένα τέτοιο γιγάντιο έργο χωρίς να υπάρχει συγχρόνως και στήριξη των λαών. Επιτυχείς τροποποίησεις και αλλαγές θα γίνουν μόνο εφόσον συμφωνεί ολόκληρη κοινωνία στο σύνολό της. Είναι αναγκαίες επίσης μεταρρυθμίσεις που θα επηρεάσουν εθνικές αποφάσεις. Οι τοπικές αρχές, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και το σώμα αυτό, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών, όλοι έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανατολική εταιρική σχέση. Γι' αυτό στηριζόμαστε στο σώμα αυτό, στο κοινοβούλιο αυτό, για να μας βοηθήσετε, να στηρίξουμε τους εταίρους μας, προκειμένου να κάνουν τις αλλαγές που επιθυμούν οι πολίτες τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you. Thank you, Minister. And, uh, Ευχαριστώ. Για τον κύριο Κέλλη και τους υπόλοιπους να πω ότι στο τέλος ε, θα δώσω μία ερώτηση κατσιδιά για ένα πολιτική ομάδα και θα δεχτώ τις μπλε κάρτες ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει η συζήτηση. Ενδεχομένως μπορεί και να μην δεχτώ μπλε κάρτες και σίγουρα δεν θα δεχτώ μπλε κάρτα από οποιονδήποτε είναι εγγεγραμμένο στη λίστα των ομιλητών. Πρώτος ομιλητής από το ΕΛΚ, ο κύριος Σάιρους Βόλσκι, για δύο λεπτά. Mrs. Vice President. Κύριε Αντιπρόεδρε, καταρχήν μην δύο φράσεις μη με τις μέτρες στο χρόνο μου. Είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιπροσωπεύεται σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Αν αυτό αποτελεί μήνυμα της σημασίας που αποδίδει η Επιτροπή σε αυτό το πρόγραμμα, λυπάμαι πάρα πολύ. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι μια πολιτική στρατηγική σημασία που έχει σχεδιαστεί πολύ καλά και μάλιστα είναι απολύτω απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι επηρεάζει την ευημερία, την ασφάλεια και την οικονομία. Ε, επίση, η βασική, βασικό στόχο είναι η ειρήνη. Χρειάζεται επίση, είναι πολύ τόσο απαραίτητη και για του γειτονέ μα, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Η ανατολική εταιρική σχέση ε, έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται, θα συνεχιστεί με, διαφορετικές, με διάφορες και ενίσχυση. Έγινε προσπάθεια να αποπροσανατολιστεί αυτή η πορεία ε, μέσω πίεση στην Ουκρανία να αρνηθεί την υπογραφή στο Βέλνιο. Στο Euromaidan όμως έδωσε μια σαφή απάντηση στις ρωσικές πιέσεις και ο λαός της Ουκρανίας είπε ότι επιθυμεί τις ευρωπαϊκές αξίες. Μετά η Ρωσία ξεκίνησε πόλεμο, ε, όμως θα αποτύχει ε, στην προσπάθεια της να σταματήσει την ανατολική εταιρική σχέση. Ε, ε, ο κανόνας λέει ότι ε, όταν δέχεσαι ε, επίθεση από ένα πουλί μην υποχωρείς. Όταν κάποιος προσπαθεί να σε σταματήσει έχεις δύο επιλογές ή να υποχωρήσεις ή να διπλασιάσεις τις προσπάθειές σου και να προχωρήσεις μπροστά. Η δεύτερη είναι η επιλογή δική μας. Διότι πρώτον αυτό επιθυμούν οι εταίροι μας. Δεύτερον διότι τα θεμελιώδη συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αξίες μας μας το επιβάλλουν. Και τρίτον, αν δεν υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και την ελευθερία στην περιοχή μας, ε, κινδυνεύει η δική μας ελευθερία, δημοκρατία και ευημερία. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαρούς Βόλσκι. Έχουμε τώρα μια μπλε κάρτα από τον κύριο Φουνσολίκα, αλλά δεν τη δέχομαι, γιατί σας είπα στην αρχή ότι θα δέχομαι μπλε κάρτες μόνο εάν ε, προέρχονται από κάποιον που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε καθυστερήσει ε, για μισή ώρα. Κύριε συνάδελφε, εσείς είστε ομιλητής για αργότερα, τώρα δεν έχει μπλε κάρτα για σας. Τέλος. Λοιπόν, ο κύριος Φλέκενστάιν από τους σοσιαλδημοκράτες παρακαλώ για δύο λεπτά. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανατολική εταιρική σχέση έχει ένα σαφή στόχο, δηλαδή επιτρέπει στους, στις γειτονικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να έχουν ένα πλαίσιο για την πολιτική και άλλη συνεργασία. Δίνει τη δυνατότητα σε ε, σχέσεις ουσίας και σε ανταλλαγές. Η ανατολική εταιρική σχέση είναι μια προσφορά για στενή συνεργασία, μια προσφορά προς ε, γειτονικές χώρες που δεν είναι ή δεν θέλουν να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα καλής συνεργασίας με την Αρμενία, με το Αζερβαϊτζάν. Τίποτα δεν εμποδίζει τη συνεργασία αυτή απλά και μόνο επειδή στις χώρες αυτές ε, έχει, ε, οι χώρες αυτές απέδειψαν ή τους απορρίφθηκε η δική τους αίτηση για ε, συμφωνία σύνδεσης. Πάντως, με πάση περιπτώσει, μπορούν αυτοί να προσανατολιστούν στις δικές μας τις αξίες. Είναι σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να αναθεωρήσει την πολιτική γειτονία και λόγω των σημαντικών προκλήσεων στην γειτονική αυτή περιοχή που τα έδειξε και ο κύριος Σαρουβόλσκι, αναφέρομαι στην Ουκρανία. παρόλα αυτά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ε, αναδιαρθρωθεί εκ βάθρων η πολιτική. Όμως η συνάντηση στη Ρήγα θα πρέπει να εκπέμψει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία της με τους ανατολικούς εταίρους θέλει να είναι όχι μόνο καλύτερη αλλά και αποτελεσματικότερη. Μεγαλύτερη αλληλεγγύη, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα συγκεκριμένα με μεμονωμένους εταίρους. Έχει έρθει η στιγμή να εστιάσουμε στα στατούτ αυτής της συνεργασίας για να ενισχυθούν οι κρατικοί θεσμοί, να υπάρξουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, βελτιωμένη περιφερειακή συνεργασία και κάτι τελευταίο. Ο πρόεδρος της Γεωργίας είπε πρόσφατα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ότι για την ε, ανατολική εταιρική σχέση είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία των χωρών και προς Δυσμάς και προς Ανατολάς. Και αυτό θα πρέπει μέσω πρόθεσμα να το έχουμε κατά νου. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο κύριος ε, Μενσμάκε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Το κείμενο που έχει ετοιμαστεί για τη διάσκεψη της Ρήγας όσον αφορά το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης είναι απογοητευτικό ως έχει. Γιατί από όλε αυτές τις μεγάλες δηλώσεις για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την στήριξη των αρχών μας δεν βλέπω τίποτα εδώ. Τίποτα. Καμία φιλοδοξία, καμία σαφή στρατηγική. Ενώ χρειάζεται τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Η πίεση της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια ήτανε σε βάρος χωρών εταίρων μας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας και ήταν τεράστια. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Δεν βλέπω όμως τίποτα για τα στρατεύματα της Ρωσίας στα ανατολικά μα σύνορα, ούτε για την παρουσία του στην Ουκρανία. Αντίθετα, η Ρωσία καλείται τελικά να καθορίσει τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Ελεύθερου εμπορίου μας με την Ουκρανία. Την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιου συναδέρφους εδώ Ήμουνα στο Κίεβο και στα ανατολικά της Ουκρανίας και είδαμε τις καταστροφικές συνέπειες της επιθετικής στάσης της Ρωσίας. Για πολλές οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στο πυρ είναι ε, φοβερό. Βλέπουμε τα βλήματα γκραντ των Ρώσων σε βάρος ε, κατοικιών στη Μαριούπολη. Οι συνέπειε είναι τεράστιε και για ολόκληρη τη χώρα. Σα προειδοποιώ λοιπόν ότι η σύγκρουση πίνει το αίμα τη χώρα, και όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Ο λαό κουράζεται και απογοητεύεται. Οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν θυσίε από τον κόσμο. Πρέπει όμω να νιώσουν ότι θα ανταμυθούν οι κόποι τους, ενώ κινδυνεύουμε να βρεθούμε απέναντι σε ητοπάθεια. Οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται ότι θα χάσουν. Συνεπώ, χρειάζεται ένα θετικό και σαφέ μήνυμα από τη Ρήγα. Πιο θετικό και πιο ε, σημαντικό από αυτό που έχουμε μέχρι τώρα στο κείμενο. Κινδυνεύουμε από τις συνέπειες. Προσοχή. Πρέπει η Ουκρανία και η Γεωργία να νιώσουν ότι μπορούμε να τους προσχεθούμε κάτι και για τις θεωρήσεις. Επόμενος εκ μέρους των φιλελευθέρων, ο κύριος Πέτρας Αουστροβίτσιους για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανατολική εταιρική σχέση ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και αποτελεί παράδειγμα της ε, πραγματικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλες τις δυσκολίες και παρόλες τις ανοιχτές επιθέσεις, η ανατολική εταιρική σχέση πρέπει να μας κάνει περήφανο σήμερα. Η ομάδα των φιλελευθέρων υποστηρίζει πλήρω την πολιτική ανατολική εσωτερική σχέση, διότι αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό κίνητρο για περαιτέρω εκδημοκρατισμό και ε, προωθεί τι ε, μεταρρυθμιστικέ διαδικασίε στου εταίρου μα στην Ανατολική Ευρώπη. Ω αποτέλεσμα, ε, τους τρεις ε, ανατολικούς εταίρους μας, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία, πρέπει να τους βάλουμε στο χάρτη της Ευρώπης γνωρίζουμε ότι πληρώνουν ένα υψηλό τίμημα ε, για την Ευρωπα... τις ευρωπαϊκές τους επιλογές. Ε, πολιτικές, στρατιωτικές, οικονομικές επιπτώσεις ε, αλλά και προπαγάνδα εναντίον τους. ξεκινήσαμε, στείλαμε ένα, μια ανοιχτή επιστολή στους αρχιούς κρατών και κυβερνήσεων ε, των, της Ευρωπαϊκής ό,τι αφορά τη δήλωση της Ρήγα αυτή η επιστολή υπογράφηκε από 98 μέλη του Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι η Σύνοδος Κορυφής της Ρήγα θα πρέπει να είναι ε, φιλόδοξη. Ε, καλούμε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρήγα να αναγνωρίσουν την, ε, τις μελλοντικές ευρωπαϊκές ε, προοπτικές των τριών αυτών χωρών. Ε, θα πρέπει να γίνουν σαφή τα κριτήρια και τα προαπαιτούμενα. Ε, και αυτό πρέπει να γίνει σήμερα, όχι αύριο. Ε, δεύτερον, στη Ρήγα θα πρέπει να χορηγηθεί ε, μια απελευθέρωση καθεστώτος θεωρήσεων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου. Η ευρωπαϊκή πολιτική ε, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία έχει αποτύχει και η ανατολική εταιρική σχέση θα ε, δώσει ε, θετικά αποτελέσματα και για σε αυτήν. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρου της Ενωμένης Αριστεράς, ο κύριος Χαλμούτο Σόλτς για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, Αύριο ξεκινάει η συνάντηση κορυφή στη Ρήγα για την Ανατολική Εταιρική Σχέση και αυτή θα είναι μια συνάντηση των αντιφάσεων. Και αυτό ήδη κάπως έχει προανακοινωθεί ε, και φαίνεται και από την πολιτική που χαράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σαρουσβολσκή, ε, σωστά το επισημάνατε ότι σήμερα λάβει δια της απουσίας της Κομισιόν. Υπάρχουν επίσης και αντιφάσεις στο περιεχόμενο. Ε, πρέπει να διερωτηθούμε τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η Μολδαβία ε, να μην μπορεί να ανατρέψει τους ε, διεφθαρμένους ολιγάρχες ε, ή πώς μπορούν άλλες άλλα κράτη να απαγορεύουν κόμματα. Στην Ουκρανία διαπιστώθηκε μια, μετά από μια έρευνα ότι ε, δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις όλες αυτές που περιμένει ο κόσμος με αγωνία από τότε, από την πλατεία του Μεϊντάν. Αυτό πρέπει να παίξει ρόλο στη Ρήγα. Και επίσης και το ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα υποφέρουν οποτεδήποτε αγνοούνται τα δικαιώματα. Μιλάμε 20% ανεργία στην Αρμενία και στη Γεωργία, στους νέους ακόμα μεγαλύτερη ανεργία ε, στη Μολδαβία, ελάχιστη απασχόληση των γυναικών. Αυτά δείχνουν ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές και όχι μόνο μια απλή αλλαγή στην αγορά. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τεθούν από εμάς, από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η ανατολική εταιρική σχέση σημαίνει κυρίως μια κοινή πολιτική και ανάπτυξη. Επόμενος ομιλητής ε, από τους ε, πράσινους, ο κύριος Τάμας ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αν υπάρχει μία κοινή πολιτική είναι, που χρειάζεται αναθεώρηση είναι η ανατολική εταιρική μας σχέση. Η ομάδα μας χαίρεται για την αναθεώρηση που ξεκίνησε ο Επίτροπος Χαν και στηρίζουμε τα συμπεράσματά του προς το παρόν. Η διαφοροποίηση είναι η λέξη κλειδί για την αναθεώρηση αυτή. Είναι κάτι λογικό και αναπόφευκτο πιστεύω όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τρεις από τις χώρες εταίρους έχουν συμφωνία σύνδεσης μαζί μας και βάσει των ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου ευθυγραμμίζονται με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε λοιπόν να τους προσφέρουμε μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή προοπτική και θα έπρεπε να τις βοηθήσουμε πρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό κόστος εξαιτίας της ευθυγράμμισης αυτής. Η αρχή περισσότερα για περισσότερα έχει νόημα μόνον εφόσον αυτό σημαίνει και λιγότερα για λιγότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα ήταν σωστό να αυξήσουμε τη, τα οικονομικά κονδύλια που είναι το 20% τώρα στα πλαίσια του More for More για τις χώρες στη σύνδεση. Και για να είμαστε αξιόπιστοι και να έχουμε αξιόπιστη πολιτική εταιρική σχέσης πρέπει να στηρίζουμε επαρκώς οικονομικά. Τα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο δεν επιτρέπει ε, πραγματική δέσμευση, ούτε φιλόδοξη πολιτική. Πρέπει να αλλάξει το νούμερο αυτό στην επόμενη αναθόρηση. Με δύο λόγια, χρειαζόμαστε αξιόπιστη δέσμευση απέναντι στους εταίρους μας και προς Νότο και προς Ανατολάς. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Καστάλντο, Φάβιο Μάσιμο Καστάλντο, για λεπτό, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πλησιάζουμε ε, σε αυτή την πολύ μεγάλη συνάντηση στην ε, ε, διάσκεψη για την Ανατολική Εταιρική Σχέση και πρέπει να πω ότι και εγώ ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι δεν παρίσταται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. πλησιάζοντας λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση κορυφής εγώ θεωρώ, εμείς θεωρούμε ότι κάποια χώρα ε, που πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης μπορεί να έχει ευρωπαϊκές προσδοκίες. Είναι όμως σαφές ότι σε πολλές από αυτές τις χώρες υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εξαρτώνται από όλα αυτά τα κονδύλια που εκταμιεύουμε ε, με τη μορφή βοήθειας και όχι να δίδονται ε, χρήματα για εξοπλισμό και για όπλα που σίγουρα αυτό δεν είναι προτεραιότητα των λαών. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σε αυτή τη συνάντηση κορφής θα προσφερθεί ευκαιρία να αναθεωρηθούν όλες αυτές οι πολιτικές. Πολύ ωραία ε, εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων ο κύριος Κόβιν Μίκε. Ε, ε, θα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια για να μην εκπλησώμεθα. Ε, κανένας δεν ξέρει ότι είναι πιο... Κανείς δεν πιστεύει ότι είναι πιο ασφαλής ένας δημοσιογράφος στη Μόσχα από ότι στο Κίεβο. Στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σκοτωθεί ένας αριθμός ε, δημοσιογράφων, τους οποίους αναφέρει ο Μιλτής, και πολλοί Ούγγροι, Μολδαβοί, Εβραίοι, Ρώσοι, από εθνικιστές Ουκρανούς. Ε, καταλαβαίνω ότι πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτούν με συμπάθεια τους εθνικιστές γιατί ο φασισμός ε, ενισχύεται. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια την οποία δεν μπορούμε να γνωρούμε. Τώρα λοιπόν ε, περνάμε σε μεμονωμένους αγορητές και το λόγο έχει ο κύριος Κρίστιαν Ταμπέρου με την Ανατολική Εταιρική Σχέση συμβαίνει κάτι παράξενο. Πριν το Βίλνιους, τον Νοέμβριο του 2013, μιλούσαμε για την αποτυχία της Συνόδου Κορυφής και υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος τώρα. Ε, γιατί κάποιοι μιλούν για μια αποτυχία ακόμα και πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής. Όμως η Σύνοδος Κορυφής του Βίλνιους δεν ήταν αποτυχία αν κάποιος κάνει τον απολογισμό ε, της κατάστασης από το 2013 μέχρι σήμερα. Ε, ε, είχαμε βήματα σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις, συμφωνίες σύνδεσης κλπ. κλπ. Προφανώς ε, η κοινωνίες οι οποίες καλύπτονται από όλη αυτή την πολιτική δεν περιμένουν απλώς ένα απολογισμό του πρόσφατου παρελθόντος αλλά και μια υπόσχεση για το μέλλον. Ένα μήνυμα όπως λέμε, μια δέσμευση σε ό,τι αφορά το μέλλον. Και νομίζω ότι εδώ είναι το ατού μας. Μπορούμε και πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον. Πρέπει να σχεδιάσουμε ε, το ευρωπαϊκό μέλλον αυτών των ε, χωρών διότι αλλιώς ε, δεν θα ε, μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ρωσική προπαγάνδα. Η Ρωσία δέχεται, αντιλαμβάνεται αυτή την εταιρική σχέση ως μια επιχείρηση αντίον της Ρωσίας. Χρειάζεται κουράγιο λοιπόν, γενναιότητα, να αναλάβουμε δεσμεύσεις για το μέλλον και θα πρέπει να είμαστε σαφείς για την ευρωπαϊκή προοπτική αυτών των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Θα ήταν κρίμα ε, σήμερα να είμαστε πιο υποχωρητικοί στις προτάσεις μας έναντι των προτάσεων που είχαμε πριν απο τρια 3-4 χρόνια στη Βαρσοβία. Voilà. Ε, der nächste ist Herr Tonino για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Η σημασία της διάσκεψης ανατολικής εταιρικής σχέσης στη Ρήγα δεν πρέπει να υποτιμηθεί επειδή αλλάζει η γεωπολιτική κατάσταση μετά την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Το κείμενο δεν είναι αρκετά ισχυρό, παρόλο που η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία στο μεταξύ έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του σύνδεσης. Αν δεν θέλουμε να τους προσφέρουμε περισσότερες ελπίδες και συμφωνώ ότι δεν πρέπει, τότε τι μένει, ποιες είναι οι, πρα... οι προπτικές ε, για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Δεν πρέπει οι χώρες αυτές εταίροι μας να νιώσουν μόνοι τους με τις πιέσεις που δέχονται και εμείς απλώς να τις κοιτάμε. Πρέπει να είναι μια ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει τη δέσμευσή της υπέρ ακριβώς αυτής της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να απαντήσουμε στο ερώτημα η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τι βαθμό μπορούν να στηρίξουν τους εταίρους τους και πόσο ευάλωτοι είναι αυτοί. Ο κύριος Κάρσκι για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε τραγική κατάσταση. η Κομισιόν, όπω είπα, λάμπει δια τη απουσία τη. Αυτή η συνάντηση κορυφή είναι καθοριστική σημασία, ίσως η πιο σημαντική ποτέ στην ιστορία ε, της ε, σχέσης μας με τις ανατολικέ χώρες. Μιλάμε για σχέσεις ε, με χώρες που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν δυσκολίε και έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προσπαθεί να σταθμίσει αντιφατικά συμφέροντα. Το κείμενο το οποίο εγκρίναμε, ή μάλλον το κείμενο που θα εγκριθεί στη συνάντηση κορφή, πρέπει να είναι ένα κείμενο ουσιαστικό. Η Ουκρανία, η Μολδαβία πρέπει να έχουν το μέλλον μπροστά τους και πρέπει να ανακοινωθεί ότι το 2016 θα καταργηθούν οι ε, βίζες ε, και για τους Ουκρανούς και για τους Μολδαβούς και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να μιλήσουμε για επιθετικότητα της Ρωσίας και προσάρτηση της Ουκρανίας. Ε, κείμενα νοθευμένα απλά θα ενθαρρύνουν τη Ρωσία για περαιτέρω επιθετικές ενέργειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ούρμας Πάιτ, για ένα λεπτό. Η πολιτική ανατολική εταιρική σχέση είναι εξαιρετικά σημαντική, αναμφίβολο αυτό. Όμως, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την ε, αυριανή συνοκορυφή, διότι θα πρέπει να κάνει κάτι πραγματικά απτό για να υποστηρίξει τις τρεις χώρες. Πλην όμως, οι ενδείξεις ε, φαίνεται ότι είναι πως ε, θα ακουστούν πολλά λόγια χωρίς πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει να θέλει να καταργήσει τις θεωρήσεις για τους Ουκρανούς. Η, η, η κοινή γνώμη στην Ουκρανία πρέπει, ε, διψάει όμως για καλά νέα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η Ουκρανία έχει μέλλον στην Ευρώπη. Ορισμένα κράτη-μέλη ε, ε, είναι ενθουσιασμένα με το μέλλον της ε, Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οκτώ χώρες δεν έχουν επικυρώσει την Συμφωνία Σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εταιρική ανατολική σχέση ήταν μια έξοχη ιδέα, όχι απλώς καλή, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατέστρεψε γιατί την εξάρτησε από την πολιτική ομοιρίας από πλευράς της Ρωσίας. 60% πληθωρισμός. Πρόβλημα με την Κεντρική Τράπεζα. Μετά τα γεγονότα της Μαϊντάν, 46 Ουκρανικές τράπεζες έχουν καταρρεύσει. Οι μισθοί κατά μέσο όρο είναι 40 ευρώ το μήνα. Οι Αμερικανοί τώρα κάνουν πίσω. Η συνάντηση μεταξύ του Κέρι, του Λαυρόφ και του Πούτιν στο Σότσι ακριβώς αυτό δείχνει. Πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν αυτή την ε, συμπεριφορά απέναντι στους Αμερικανούς. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπρόνις Ρόπε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ρωσία ε, φαίνεται να απειλεί έμεσα ότι αυτό που σημαίνει στην Ουκρανία μπορεί να συμβεί και σε άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ε, απειλή, με οικονομικές κυρώσεις και με άλλες κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά σε αυτό, σε αυτές τις απειλές θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ισχυρή. Θα πρέπει να δώσουμε πραγματική στήριξη στις χώρες της εταιρική σχέσης. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και θα πρέπει να ενημερώσουμε αυτές τις χώρες καλύτερα για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το Κοινοβούλιο και για την ομοθετική διαδικασία που ακολουθούμε. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και καλύτερα την εργασία των δημοσιογράφων αυτών των χωρών εδώ, στο Στασβούρο και στις Βρυξέλλες. Ε, θα πρέπει να προβούμε σε ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, ε, ενημέρωσης, ιδιαίτερα με τις χώρες της ε, Ανατολικής Εθερικής Σχέσης. Θα πρέπει να ακούσουμε ποιες είναι οι πραγματικές ελπίδες των πολιτών και να επενδύσουμε ιδεολογικά σε αυτές τις χώρες. Η σύνοση κορυφή γίνεται αύριο. Ε, μιλάμε σαν να έχουμε ήδη πετύχει, συμπεριλαμβανομένων και των σχέσεων με την Ουκρανία παράξενος ο ορισμός της επιτυχίας αν δει κανείς την κατάσταση επικρατεί στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Ε, συμπάσχουμε με, το λαό εκεί. Ή το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τίνει να επεκτείνει την εξουσία της ε, και το πεδίο της σε όλο και περισσότερες χώρες χωρίς όριο. γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η σχέση της ε, Ρωσίας, ε, η οποία αμφισβητεί την ειρήνη και τη θέτει σε κίνδυνο. Ε, στο Star Trek υπάρχει ένας εχθρός που ονομάζεται The Bog και προσπαθεί να κάνει όλους οι υπόλοιπους ίδιους με αυτόν και είναι ο μόνος λόγος ύπαρξής του αυτός όσο πιο πολύ είμαι στο κοινοβούλιο, τόσο πιο πολύ βλέπω ότι γινόμαστε Star Trek. Ε, να επηρεάζουμε όλο και περισσότερο, να δεσπόζουμε όλο και περισσότερο, να επεκτηνόμαστε όλο και περισσότερο. Ας κάνουμε μια παύση και ας σκεφτούμε λίγο. Απογοητεύομαι, αποκαρδιώνομαι όταν ακούω τι γίνεται και ελπίζω δεν θα βγει τίποτα κακό από αυτή τη σύνοκορυφή. Ε, Κύριε Γιουρίκ, είδα ότι θέλετε μπλε κάρτα, αλλά σας βλέπω στον κατάλογο μου των ομιλητών, γι' αυτό λοιπόν δεν σας εγκρίνω την μπλε κάρτα, μπορείτε να μιλήσετε αργότερα. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σορτεμπάλτσοφ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η ανατολική εταιρική σχέση είναι κάτι το οποίο εμείς ε, δρομολογήσαμε εν μέρη για να διαφοροποιηθούμε από τις ενέργειες της ε, Ρωσίας. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί και όταν υπάρχουν κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες που δεν λειτουργούν σωστά πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Ένα πράγμα είναι σαφές. Υπάρχει υποστήριξη εκ μέρους των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχουν μέτρα που έχουν ληφθεί όμως ε, στις χώρες αυτές ε, καταπιέζονται και οι μειονότητες ε, και δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους σε αυτές τις χώρες ε, συμβαίνουν πάρα πολλά τα οποία αντιβαίνουν στα δικά μας τα δικαιώματα. Αν λοιπόν θέλει κανείς να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ να μιλήσουμε καθαρά. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Αντρέ Μπλένκοβιτς για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ε, ευχαριστώ πολύ αυτή η συζήτηση για την τέταρτη συνάντηση κορυφής Ανατολική εταιρικής σχέσης του θα λάβει η χώρα στη Ρήγα είναι πολύ σημαντική για την αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα ε, προς τις ε, πέντε χώρες που συμμετέχουν περισσότερο. Δεν μιλάω για τη Λευκορωσία. Αυτή έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Τα μήνυματα αυτά διαφέρουν κατά πολύ από αυτά που στείλαμε στο Vilnius. Αυτό που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι θέλουμε να τις επιβραβεύσουμε για τον δρόμο που ακολουθούν ε, κυρίως την Γεωργία και τη Μολδαβία. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουν τις προσπάθειες προσπάθειές να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα μέτρα που μπορούν. Η οικονομική αρρωγή, η δημιουργία ε, θεσμών, ε, δικαστική βοήθεια κυρίως στον αγώνα κατά της διαφθοράς, αυτά θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες ε, στις πολιτικές μας τα μηνύματα που στέλνουμε στους πολίτες αυτών των κρατών, κυρίως όσον αφορά την απελευθέρωση του καθεστώτος της θεώρησης, αυτά τα μηνύματα είναι πολύ σημαντικά για την κοινή γνώμη. Ε, κατά τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικό, επειδή δώσαμε άλλα μηνύματα, είναι σημαντικό να μην τους απογοητεύσουμε και πρέπει να καταστήσουμε σαφές και στις γειτονικέ χώρες ότι όλοι αυτοί οι εταίροι έχουν σαφώς το δικαίωμα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μποστινάρου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, από την τελευταία συνάντηση κορυφή στο Βίλνιους έχουν αλλάξει πάρα πολλά ε, στη σχέση μας ε, με τους εταίρους. Κυρίως αυτοί που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί αντιμετωπίζουν τεράστια εξωτερική πίεση. Στην Ουκρανία μάλιστα αυτή η εξωτερική πίεση τι είναι, είναι πόλεμος υπάρχουν τα στρατεύματα των Ρώσων που περνάνε τις ε, διακοπές τους στην Ανατολική Ουκρανία με ένοπλα τεθωρακισμένα οι χώρες ε, της Ανατολική εταιρικής σχέσης ε, θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι εταίροι και να ενισχυθούν στις προσπάθειές τους για μεταρρυθμίσεις, αλλά επίσης να αναγνωρίζουμε και την πρόοδο οποτεδήποτε αυτή λαμβάνει η χώρα. Αν δεν υπάρχουν υψηπετείς φιλοδοξίες στη Ρήγα, αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες ε, στην Ευρώπη, κυρίως στην ανατολική της πλευρά. Απευθύνομαι και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι από τη Ρήγα θα θετικό μήνυμα προς τους ανατολικούς μας εταίρους. Εγώ δύο λεπτά έχω κυρία Πρόεδρε, όχι ένα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να καταπνίξει τις προσδοκίες ε, των εταίρων μας και των πολιτών τους ε, του αντίον να κάνει το αντίθετο. Να δείξει ότι είναι ανοιχτή η Ευρωπαϊκή Οδός περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν να τους προσφέρει τη δυνατότητα ε, να ανταπεξέλθουν στην ισχυρή πίεση της ρωσικής προπαγάνδας. Πρέπει να γίνει ένα μεγάλο βήμα, δηλαδή απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για την Ουκρανία και τη Γεωργία. Ας μην δώσουμε τίποτα άλλο, ας δώσουμε κάτι που μπορούμε να το δώσουμε και με βάση τις προσπάθειες που κατέβαλαν αυτές οι χώρες. Είναι το πρώτο σημαντικό ε, μήνυμα ότι το μέλλον τους είναι στην Ευρώπη, πρέπει να συνεχίσουν να παλεύουν γι' αυτό. Και θέλω να σας πω ότι ε, και εγώ στηρίζω την επιστολή που έστειλε ο συνάδελφός μας, ο κύριος Οστρεβίτσιος. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Κοσματοφστόφσκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση και η Σύνοδος Κορυφής είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να παριστάνει ότι έχει μια τέτοια πολιτική, να την κάνει πράξη. Κοιτάξτε τι γίνεται με την Ουκρανία. Εάν η στρατιωτική ρωσική δράση δεν αποτελεί αρκετό κίνητρο για μας για να αντιδράσουμε, να κάνουμε κάτι για τους εταίρους μας στην ανατολική εταιρική σχέση, τότε ποιος θα το κάνει. Η Ουκρανία είναι πάνω-πάνω στην ατζέντα. Υπάρχει χάος, φόβος για τόχευση Καταστρέφεται η χώρα αυτή, καταστρέφεται και η ίδια η αρχιτεκτονική ασφάλεια στην, ε, στις πόρτες μας. Η οικονομική αρρωγή λοιπόν είναι αναγκαίο προς τους θεσμούς της Ουκρανίας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής. Και το ίδιο ισχύει και για τη Γεωργία και για τη Μολδαβία. Η δύναμη της Ρωσίας είναι δικιά μας η δυναμία. Και αντίστροφα. Πρέπει να είμαστε σταθεροί, αλλά βλέπω ότι η Επιτροπή δεν κάνει καν τον κόπο να είναι εδώ. Ο κύριος Ιβο Μπάγγελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι θα μου αφαιρέσετε το λόγο, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να πει κάποιος κάτι περίπλοκο σύντομα και συνοπτικά. Η ε, Ανατολική Εταιρική Σχέση και η Ένωση για τη Μεσόγειο αποτελούν καινοτομίε τη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ε, που δεν είχαν εμφανίσει επιτυχίε για πολύ καιρό. Γι' αυτό το λόγο μιλούμε σήμερα για την ανατολική εταιρική σχέση και την ανάγκη αναθεώρηση τόσο αυτή όσο και τη Ένωση για τη Μεσόγειο που έχουν γίνει όμοιροι διμερών εκρεμών ε, θεμάτων και αντικρουόμενων γεωστρατηγικών συμφερόντων. Ε, όμως το κοινό χώρο αξιών μα ε, πρέπει να διευρυνθεί και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες σε αυτή τη μεριά του κόσμου, σε αυτή την περιοχή. Είμαι πεπισμένο ότι αν βλέπαμε με αυτόν τον τρόπο ε, τις εταιρικέ σχέσεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε λάβει χώρα. Θα συνεχίσω μια επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Und nun Herr Javier Javier Η ανατολική εταιρική σχέση, όπως ε, σχεδιάζεται στη Ρήγα, δεν μα αρέσει. Οι συμφωνία σύνδεση, οι ζώνε ελεύθερων συνταραγών ε, είναι όπλα πολιτικού ελέγχου ε, με ανισότιμε οικονομικέ σχέσει. Εμεί, οι χώρε του Νότου γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό περισσότερο χρέο από βιομηχάνηση και ε, ε, πιο ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Ε, έχει μετακινηθεί με παράνομο τρόπο η εξουσία, έχει δημιουργηθεί, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες πολέμου κλπ. με αυτή την πολιτική. Και το ΝΑΤΟ είναι ακόμα πιο επιθετικό. Και μιλάμε για ένα ευρυδικό πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό πιο πολύ ε, χρησιμοποιείται για τις σχέσεις Ελλάδας με τη Ρωσία παρά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, το, τελικά όλα εξαρτώνται από τις επιθυμίες ε, της, των ΗΠΑ και σίγουρα αυτή η πολιτική δεν είναι πολιτική ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. και η κυρία Τατιάνα Στανόκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι δεν συμμερίζομαι την ε, αισιοδοξία του προαλήσαντος. Η ανατολική εταιρική σχέση είναι παγίδα για συγκρούσεις και η μόνη δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να παρεμποδίσει την επιδείνωση των σχέσεων με τη Ρωσία και να σταματήσει την πίεση που ασκείται στους λαούς ε, που βρίσκονται στην πλευρά αυτή, στην ανατολική πλευρά. Ε, είναι και θέμα ερμηνείας γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει μια επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία είναι το δηλητήριο που προέκυψε από αυτή τη διαστεύρωση. Σήμερα, 40 χρόνια μετά την θέσπιση της τελικής πράξης του Ελσίνκη, είναι πηγόντως απαραίτητο να υπάρξει μια νέα συνδιάσκεψη για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αλλά και αυτό ε, αν δεν το κάνουν οι εταίροι, τότε θα το κάνουν οι κοινωνίες των πολιτών. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενώνει και όχι να διαιρεί. Και τώρα λοιπόν ο κύριος Σαφχάουζ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία εκπρόσωπη της κυρίας Μογκερίνη, τις παραπονές στη Συνόδου Κορυφή στη Ρήγα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό Τη Ανατολική εταιρική σχέση. Καμία υπόσχεση που είχαμε κάνει πριν στο ψυχρό πόλεμο δεν έγινε πραγματικότητα. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα ενώσουμε την Ανατολή και τη Δύση σε μια ανεξάρτητη Ευρώπη. Ενώ η πολιτική μας, ενώ ξέρουμε ότι κάποιες χώρες αποτελούν γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δύση, τελικά είναι οι λαοί οι οποίοι συγκρούονται μεταξύ τους. Και όλα αυτά για τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για τη Σερβία, για τη Γεωργία, είτε για την Ουκρανία, για να αναφερθώ στι χώρε σύγκρουση. Σίγουρα έχουμε ξεπεράσει τα 10.000 θύματα στην Ουκρανία. Και άλλε συγκρούσει θα λάβουν χώρα όσο εμεί στηρίζουμε μια πολεμική πολιτική αντίσταση στο ΝΑΤΟ κατά των Ευρωπαίων. Είμαστε υπέρ στον κύριο Κέρι υπέρ μιας ρεαλιστικής πολιτικής που θέλει και η εκπροσωπός μας. Μην έχουμε δύο μέτρα και σταθμά και πρέπει να έχουμε μια νέα πολιτική, μια ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κέλλαμ για 1,5 λεπτό. Η συνόδος κορυφής της Ρίγα δεν θα πρέπει να γίνει ε, σύνοδος ελάχιστων πολιτικών δεσμεύσεων όπως μερικοί προβλέπουν. Ε, ξέρω ότι πολλοί δεν θέλουν να δώσουν υποσχέσεις. Άλλοι όμως πιστεύουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να σωθεί αυτή η περιοχή. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει προσήλωση και αφοσίωση στους ανατολικούς εταίρους ε, αυτός είναι ο δρόμος προς τη δημοκρατία. Μ' αρέσει η δήλωση του Προέδρου της Λετωνίας ότι ε, ε, χρειαζόμαστε μια ε, πραγματική ανάληψη ευθυνών. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Είμαι ένας από αυτούς που έχουν υποβάλει την επιστολή προς την ε, Σύνοκορυφή της Ρήγα να υπενθυμίσω λοιπόν, να επαναλάβω την έκκληση του χρόνου να έχουμε ένα καθεστώς ε, χωρίς θεωρήσεις για την Ουκρανία και τη Γεωργία και μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική και για τις τρεις χώρες που το επιθυμούν. Η υποχρέωση μας άλλωστε είναι να εγγυηθούμε ότι αυτές οι χώρες θα επιλέξουν ελεύθερα το μέλλον τους. Η προσέγγιση μας θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ε, ανά χώρα, αλλά το μήνυμα θα πρέπει να είναι ότι δεν θα πρέπει να γίνουμε πιο ήπιοι στις δεσμεύσεις μας, δεν θα πρέπει να τους απογοητεύσουμε, θα πρέπει να τους καλωσορίσουμε το συντομότερο στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ευχαριστώ. Επόμενος μιλητής, ο κύριος Ανδρέας Μαμικίνης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το σημαντικότερο καθήκον αυτής της ε, συνάντησης κορφής είναι να απαντήσει στην ερώτηση κατά πόσον ε, θα υπάρξει μεταρρύθμιση στο περιεχόμενο της εταιρική σχέση ή κατά πόσον αυτή ε, θα πεθάνει. Δεν είδαμε να λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις και δεν είναι σαφές ε, γιατί ε, δεν έχουν καταργηθεί οι θεωρήσεις με τη γεωργία που έχει καλύψει όλες τις προϋποθέσεις. Νομίζω ότι η Κομισιόν πρέπει να λάβει μια θετική απόφαση, αλλά γιατί δεν ελήφθη αυτή στο παρελθόν. Είναι θέμα προσέγγισης. Δεν βλέπουμε ότι είμαστε επιρμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί ε, να παίζει το ρόλο του μεγάλου αδελφού. Αυτό είναι λάθος. Ε, η άλλη πλευρά επιθυμεί να ε, μιλούμε ως ίση προς Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί το πρόγραμμα της Ανατολικής Τερικής Σχέσης. Ευχαριστώ. Επόμενος ο μιλτής, ο κύριος Μανακιούρεκ, επίσης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ενισχύοντας την ανεξαρτησία των χωρών που προέκυψαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση δίνουμε ουσία και περιεχόμενο στη συνεργασία μας. Μιλήσαμε, κάποιος μίλησε για ρεαλισμό και σεβασμό της σφαίρας συμφερόντων και επιρροής της Ρωσίας. Αν μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα ε, υποσκάπτουμε τον ηθικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κηρύττουμε τις αξίες μας και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτές οι χώρες, κυρίως η Ουκρανία και η Γεωργία, θέλουν να φέρουν σε μας και τις δικές τους αξίες που μπορούν να μας ωφελήσουν. Ο, η χριστιανοσύνη επιβίωσε για αιώνες. Αυτό το λάβαμε υπόψη μας ε, στις, ε, στα ψηφίσματά μας. Ε, ο μιλήσω και ο Στετίνα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση κορυφής στη Ρήγα θα είναι μια ευκαιρία για να διαφοροποιηθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις έξι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Από την άλλη βέβαια πρέπει να υπάρχει μια ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις χώρες αυτές. Ας δούμε ποιος είναι ο κοινό παρανομαστής. Τρεις βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, Αρμενία κατά το Αζερβαϊτζάν, Ουκρανία με τη Ρωσία. Ε, τρεις χώρες είναι εν μέρη υποκατοχή, Γεωργία, Νότια Οσετία και Απχαζία, Μολδαβία, Υπερδνηστερία, Ουκρανία, Κρυμαία. Η έκτη χώρα είναι η Λευκορωσία που δεν κρύβει τις ανησυχίες της για την ασφάλειά της. Ο κοινό παρονομαστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η, βίαιη και η υπεριαλιστική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Απευθύνομαι στον Επίτροπο Χαν να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Η Ρωσία έχει κηρύξει υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης και υβριδικό πόλεμο κατά των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που προσπάθησαν να αποτινάξουν τον αυταρχικό ε, ζυγό της Ρωσίας ε, πρέπει λοιπόν επιτέλους να πούμε την αλήθεια για τη Ρωσία. Η Ρωσία για άλλη μια φορά έχει γίνει η αυτοκρατορία του κακού και επηρεάζει αρνητικά κυρίως τις έξι χώρες της δικής μας ανατολικής εταιρικής σχέσης. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Σάνι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου μίλησε εκ μέρους και της Επιτροπής και νομίζω ότι μας έδωσε καλά νέα. Τι περιμένουμε λοιπόν από τη Συνοδοκορυφή της Ρήγα. Περιμένουμε να πάρουμε και πάλι τα πράγματα στα χέρια μας, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές που είναι σε κατάσταση αποσταθεροποίησης. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε συγχρόνως και τα προβλήματα τα οποία παραμένουν. Κάποιοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ουκρανία για παράδειγμα, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι μια χώρα που τις επιτέθηκαν και βρίσκεται ένα κομμάτι της υποκατοχή. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική για τη χώρα αυτή. Συνεπώς πρέπει να προετοιμαστούμε για την σύνοδο αυτή Πρέπει να προετοιμαστούμε για τέτοιες κρίσεις και για τέτοια προβλήματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν στα σύνορά μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε άλλες μεγάλες χώρες να έχουν την πρώτη θέση στο χωρό. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες εμείς ήδη. Ο κύριος Ντέβιτ Μαγκέλης για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, υπάρχει ένα σαφές ε, πολιτικό μήνυμα, αυτό θα πρέπει να βγει από τη Ρήγα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τους εταίρους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, με συνέπεια μάλιστα και επειδή υπήρξαν κάποια πράγματα που άκουσα σήμερα και με ξένησαν, λέχτησαν τόσο από την ακραριστερά όσο και από την ακραδεξιά, θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω ότι η ανατολική εταιρική σχέση δεν σημαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Δεν πρόκειται για το είτε είτε, αλλά πρόκειται για το και το ένα και το άλλο. Η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση δεν στρέφεται κατά κανενός, ούτε κατά της Ρωσίας. Για τις χώρες αυτές, ε, οι χώρες αυτές μόνες τους θα αποφασίσουν κατά πόσο επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν, είναι, δεν επιθυμούν όλες οι χώρες να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ίδια ταχύτητα. Γι' αυτό λοιπόν ε, στη συνεργασία με τις χώρες αυτές θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να συνεχίσει να προβάλλει αξίες όπως δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να είναι ένα θέμα της επικείμενης συνάντησης κορυφής στη Ρήγα. Ευχαριστούμε πολύ η ε, κυρία Κλεμούτη είναι στον κατάλογό μου για ένα λεπτό, αλλά δεν νομίζω ότι βρίσκεται στην αίθουσα. Άρα δηλαδή, επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Έντουαρτ Κούκαν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τρέχουσα κατάσταση στα ανατολικά των συνόρων μας μοιάζει με επιστροφή στις παλιές πολιτικές ε, ε, μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ε, η συνεργασία μας ε, με αυτές τις χώρες είναι πολύ σημαντικό πλαίσιο. Ε, στόχος είναι, μια πιο, είναι πιο δημοκρατική και πιο ευημερής και πιο ενταγμένοι γείτονες. Θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτές τις βασικές αρχές. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε πολιτικό κεφάλαιο στους γειτονές μας. Θα πρέπει να ε, συμμετέχουμε όλοι, δίνοντας ένα κοινό, ισχυρό μήνυμα μέσω της Συνόδου Η πολιτική γειτονία μας θα πρέπει να έχει ε, μεγαλύτερη, καλύτερη, πιο ισχυρή πολιτική κατεύθυνση. Θα πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένο ε, προσανατολισμό και προοπτικές στους γειτονές μας και θα πρέπει οι πράξεις να ακολουθούν τις ιδέες μας και τα λόγια μας. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μήνυμα από εμά τώρα, περισσότερο από ποτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κριστέα, ένα λεπτό. Όπως συζητάμε, ετοιμάζονται αλλαγές στα ανατολικά μας. Σε μερικά χρόνια θα πρέπει να μπορούμε να κοιτάμε πίσω με την πεποίθηση ότι κάναμε το σωστό και ανταποκριθήκαμε σωστά στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανατολική Ευρώπη. Θα αναφερθώ στη φιλοδοξία και στις προπτικές. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στις χώρες εκείνες που έχουν πραγματικές ευρωπαϊκέ φιλοδοξίε που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό δρόμο. Φυσικά και πρέπει να γίνουν περισσότερα και τα λόγια δεν είναι τόσο αξιόπιστα όσο απτέ πράξει. Όμως πρέπει να δώσουμε στη Μολδαβία, στη Γεωργία και στην Ουκρανία κάποια δείγματα για το ότι το μέλλον τους είναι μαζί μας. Εφόσον βέβαια τηρούν τις υποχρεώσεις τους και δείξουν πραγματική δέσμευση στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης. Πρέπει να μπορούν να δούνε φως στο τέλος του τούνελ. Πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας σαν σοβαρές υποψήφιες χώρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Ζορογεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι η πολιτική μας προς τους εταίρους μας της ανατολικής εταιρικής σχέσης ήταν πάντα κάτι το αφελές, κάτι χωρίς συνοχή. Ειλικρινά, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Τα τελευταία όμως πέντε χρόνια έχουμε προδεύσει. Εξακολουθούμε να μην ε, αντιμετωπίζουμε με συνοχή την κατάσταση. Δεν καταφέρουμε πάντα να προσφέρουμε αυτό το οποίο θα έπρεπε να προσφέρουμε, αλλά λίγο πολύ είμαστε στο σωστό δρόμο. Τώρα, θέλω να τονίσω εδώ ότι στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης πρέπει να διαφοροποιήσουμε τους εταίρους μας. Αυτό που προσφέρουμε στους εταίρους μας πρέπει να βασίζεται στις διαφορές που υπάρχουν αναπόφευκτα μεταξύ τους, δεδομένου ότι πρόκειται για έξι διαφορετικές χώρες. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, μερικές φορές και διαφορές νοτροπίας μεταξύ τους ή πολιτισμικές. Θέλω λοιπόν να απαντήσω εδώ σε κάποιες επικρίσεις που ακούστηκαν από την είπα το εκπρόσωπο που πολύ συχνά έρχεται εδώ στο σώμα και υπάρχει φαντάζομαι κάποιος λόγος για τον οποίο δεν βρίσκεται εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στρογεύσκη. Ε, τα είχατε άλλα 20 δευτερόλεπτα, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστούμε πολύ που τελειώσετε νωρίτερα. Και τώρα ε, για ένα λεπτό ε, επόμενος ομιλητής ο κύριος Προντσουλίκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Λουκάστεβιτς είπε ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρουμε μια ουσιαστική σχέση σε αυτές τις χώρες. Δυστυχώς όμως προσφέρουμε λιγότερα από τις προσδοκίες τους. Κατ' ουσίαν όπιστο χωρούμε σε σχέση με την ανατολική ε, τερική σχέση που αποφασίστηκε στο Βίλνιους. Κυρίε και κύριοι, οι χώρες αυτές χρειάζονται μια ουσιαστική ευρωπαϊκή προεπτική. Αυτό επιθυμούν και δυστυχώς ε, σε αυτή την συνάντηση που θα ξεκινήσει αύριο αυτές τις τρεις χώρες ε, τις μετατρέπουμε σε ένα είδο χώρες μαξιλάρι εισαγωγικά ε, είναι ένα βήμα προς τα πίσω είναι ένα είδος παραχώρησης προς τη Ρωσία. Συμφωνώ με το Συμβούλιο ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη των συντομότερων δυνατών να επικυρώσουν τη συμφωνία σύνδεσης, να υπάρχουν ουσιαστικές εμπορικές ανταλλαγές με την ε, Γεωργία, την Ουκρανία. Αυτές είναι απαραίτητες για να ενισχυθεί η πολιτική συνεργασία και η οικονομική ολοκλήρωση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Επόμενη για 1,5 λεπτό η κυρία Ντουμπράφκα Σουίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντιμετωπίζουμε μια καινούρια γεωπολιτική κατάσταση σήμερα σε σχέση με αυτήν που επικρατούσε πριν τη σύμμοκορφη του 2013. Ε, η κατάσταση άλλαξε με χρήση βίας. Οι χώρες για τις οποίες ε, ομιλούμε βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση μεταξύ τους. Τρεις από αυτές είναι παρόμοιες, ε, βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, αλλά οι άλλες είναι σε διαφορετική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ε, έχουν επέλθει πολλές αλλαγές από το 2013 και μετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθεί στην ίδια οδό, πρέπει να ακούσουμε τους εταίρους μας. Όπως είπε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου, θα πρέπει να τους ε, προσφέρουμε μια πλήρη εταιρική σχέση, μια σοβαρή εταιρική σχέση. Είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν κατάφερε να μας αποπροσανατολίσει και γι' αυτό λόγο εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ενδεχομένω τη Ρωσία εχθρό, αλλά σίγουρα είναι αντίπαλος. Το γεγονός είναι ότι οι πολίτες αυτών των κρατών περιμένουν αλλαγές και γι' αυτό το λόγο πρέπει να επιμείνουμε. Θα πρέπει να τους προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική και οι συμφωνίες ε, σύνδεσης ε, υπογράφηκαν, έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν καρπούς, ο βασικός μας στόχος όμως είναι η ειρήνη. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επιμείνουμε. Όχι μόνο αλληλεγγύη αλλά και ε, στήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μιχαήλ Κάλε για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα αποτέλεσμα σε αυτή τη συνάντηση το οποίο θα ενθαρρύνει τους ανατολικούς μας εταίρους. Να τους ενθαρρύνει όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική στο βαθμό βέβαια που το επιθυμούν. Έχω την εντύπωση ότι ορισμένε από αυτές τις χώρες δεν επιθυμούν αυτή την προοπτική ε, και εμείς δεν θα, το, δεν τους το επιβάλλουμε. Η προοπτική πρέπει να είναι δημοκρατία, ελευθερία, κράτος δικαίου σε αυτή την πλευρά της Ευρώπη Γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η ρωσική Πολύ συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ε, πέσουμε και πίσω από την απόφαση του Βίλνιους ε, το 2013. Πρέπει να καταστήσουμε σαφή τη ρωσική επιθετικότητα κυρίως στους ανθρώπους στην Ουκρανία αλλά και στη Γεωργία ε, σαφώς και οφείλουμε να εκταμιεύσουμε εκατομμύρια προς την Ουκρανία αλλά και κάτι άλλο που δεν μας στοιχίζει τίποτα. Δηλαδή να τους καταστήσουμε σαφή τα συναισθήματά μας ε, κατανόησης και συμπάθειας ε, και αυτό σημαίνει γιατί όχι να καταργήσουμε τις ε, θεωρήσεις. Αυτό αναφέρεται και σε μια επιστολή που έστειλαν κάποιοι συνάδελφοι. Νομίζω λοιπόν ότι με την ευκαιρία αυτή τη συνάντηση κορυφή θα έχουμε τη δυνατότητα να τους προσφέρουμε αυτή τη συγκεκριμένη προοπτική έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα ότι είναι και αυτή ένα κομμάτι της ελεύθερης Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λέσλο Τόκιος για ένα λεπτό παρακαλώ, είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, η στρατιωτική κρίση Ουκρανίας και Ρωσίας έχει δημιουργήσει μια νέα γεωπολιτική κατάσταση για τις χώρες που ανήκουν στην ανατολική εταιρική σχέση. Η Σύνοδος της Ρήγας θα λάβει χώρα σε αυτό το πλαίσιο που είναι γεμάτο προκλήσεις και παρουσιάζει πολλά προβλήματα, διότι είναι και πολύ περίπλοκο. Η συνάντηση αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να στείλει ένα θετικό και ενθαρρυντικό μήνυμα στους εταίρους μας παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία της Σύνδεσης. Με αναφέρομαι στην Μολδαβία, στη Γεωργία μεταξύ άλλων, χώρες που είναι αρκετά διαιρεμένες. Θα πρέπει να βρούμε μια πολιτική λύση στην κρίση Ουκρανίας-Ρωσίας και στην κρίση Ευρώπης και Ρωσίας για να αποφευχθεί ο πόλεμος και να επιτευχθεί η ασφάλεια και η σταθεροποίηση της περιοχής. Θα πρέπει να στηρίξουμε την εταιρική ανατολική σχέση χαράσσοντας σαφείς γραμμές, περιχαρακώνοντας το πλαίσιο για την προσχώρηση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνοντας σε αυτές τις χώρες προοπτική. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπόνι για ένα λεπτό. Είναι πολλές οι προσδοκίες ε, της Συνόδου ε, της Ρήγας λόγω των, της επιθετικής στάσης της Ρωσίας θα μας άρεσε να έχουμε πιο ισχυρά, πιο έντονα επιτεύγματα. Θεωρώ ότι μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος, έστω και μικρή. Μιλούμε για τη διαδικασία προσχώρησης τριών ε, χωρών μελών. Προσπαθούμε να καθορίσουμε νέους όρους για την πολιτική γειτονία, για την ανάπτυξη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, για την εδραίωση του κράτους δικαίου μεταξύ άλλων. Στηρίζουμε μεταρρυθμίσεις ζωτικής σημασίας Είμαστε σε καλό δρόμο και με τις υπόλοιπες χώρες, Αρμενία, Αζερβατζάν και δεν ξέρω αν εκεί εντάσσεται και Λευκορωσία. Το πιο σημαντικό είναι να σταλεί ένα θετικό μήνυμα στις κοινωνίες, στους λαούς, ότι δηλαδή ε, παρά το ότι υπάρχουν απειλές από την Ρωσία είναι χώρες δικαιούχοι σε πάρα πολλά πεδία. Π.χ. πλήρη απελευθέρωση της έκδοσης ε, θεωρήσεων, της έκδοσης θεωρήσεων για Ουκρανία και Γεωργία προοπτική ε, προσέγγισης και προσχώρησης στο απότατο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε. Κύριε Γκρίσπ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πριν ε, τη Σύνοδο για την Ανατολική Γειτονία, Σκεφτόμασταν τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να έχουμε πετύχει παραπάνω, αν ε, υπήρχε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα μεταξύ μα. Αυτή η πρωτοβουλία δεν ήταν ε, ειδικά κατά κάποιου, ειδικά κατά της Ρωσίας, όπως φαίνεται ότι κάποιοι υπονοούν. Η εταιρική σχέση αυτή είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ έξι κρατών εταίρων με διαφορετικές ε, ικανότητες, με διαφορετικές φιλοδοξίε. Ω τώρα έχουμε πετύχει πολλές ε, συμφωνίες ε, εταιρική σχέσης με την Ουκρανία, την Γεωργία και τη Μολδαβία και άλλα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα ταμεία για την ανατολική, για την σχέση. Είναι διαφορετικέ λοιπόν οι φιλοδοξίε και θα πρέπει ανάλογα διαφορετικέ να είναι και οι προσδοκίε μα. Καλώ ορίζω το γεγονό ότι η Μολδαβία, η Γεωργία και η Μολδαβία έχουν επιλέξει το ευρωπαϊκό μονοπάτι. Ευχαριστώ κύριε Σκέλη. Σα ευχαριστώ. Καταρχά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον, την Πρόεδρο που διευκρίνησαν τα πράγματα για τι μπλε κάρτε και έτσι ήταν πολύ δομημένη και διαρθρωμένη η συζήτηση. Ευχαριστώ. Κατά δεύτερον, εδώ στο Κοινοβούλιο είμαι εδώ και έξι χρόνια. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που βλέπω το Συμβούλιο εδώ. Σε κάποιες φορές ε, ε ασκούνται κριτικέ ε, για την παρουσία του Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι εδώ πέρα σε μια τέτοια συζήτηση του Συμβουλίου. Αλλά η αδράνειά τους θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη δική μας αποφασιστικότητα προκειμένου να υπάρχει επιτυχία στα αποτελέσματα στη Ρήγα. Και πάνω απ' όλα, νομίζω ότι οι χώρε αυτές έχουν καταδείξει με μεγάλα γενναιότητα ότι έχουν το ρητό East is και West is best, ότι η Δύση είναι καλύτερη επιλογή για αυτούς. Και σε ό,τι αφορά την κατάσταση θεωρήσεων το 2016 είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και θα ενθαρρύνει τους πολίτες και γι' αυτό λοιπόν θα ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι και θα σεβαστούμε τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες τους. Ευχαριστώ. Τελείωσε ο γύρος των παρεμβάσεων στο ΚΑΣΤΙΑΙ και ξεκινάμε τον κύριο Χέτμαν πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η ε, Σύνοδος Κορυφής για την Εταιρική Γυτνίαση ε, είναι η λιδία λίθος ε, όλων των πρωτοβουλειών που συζητούμε και γι' αυτό περιμένουμε πολλά ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ημερήσιας διατάξεως είναι η συνεργασία για τον ασφαλή εφοδιασμό σε ενέργεια, για τις διασυνδέσεις. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε δοκιμές αντοχής, αναλύοντας ενδεχόμενες συνέπειες ε, του σταματήματος της πάυσης της διακοπής της ροής φυσικού αερίου από Ρωσία προς μας και απεδείχθη ότι καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να μειώσουν τα προβλήματα να αυτά διαφανούν. Έχουμε μια αστάθεια στον κόσμο σήμερα και θα πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος τον ασφαλή εφοδιασμό σε ενέργεια. Γι' αυτό καλωσορίζουμε οποιαδήποτε πρόταση που αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια και αναπτύσσει τις ε, διασυνδέσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, δράτω με της ευκαιρίας για τη συζήτηση για την ανατολική εταιρική σχέση για να αναφερθώ σε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά στους ελληνικούς πληθυσμούς που κατοικούν στη Γεωργία. Σε μια περιοχή όπου παραδοσιακά πριν από αρκετές δεκαετίες κατοικούσαν πάνω από 150.000 Έλληνες, οι οποίοι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης οι περισσότεροι ήρθαν στην Ελλάδα. Παραμένουν όμως εκεί 15.000 Έλληνες το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι μετά την αποχώρησή τους από την γεωργία όπου ήταν και πολίτες της γεωργίας άφησαν τα σπίτια τους τα οποία όμως ήταν δικά τους ήταν στη διοκτησία τους. ταυτόχρονα όμως μετά την αποχώρησή τους έγινε μια παράνομη κατάληψη των ίδιων των σπιτιών τους. παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει συνεχίζει αυτή η παράνομη κατάληψη των σπιτιών των ελλήνων πολιτών και οι αρχές της γεωργίας δεν παίρνουν μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των ελλήνων πολιτών. ζητούμε λοιπόν να ληφθεί αυτό σοβαρά υπόψη από την προεδρία αυτή τη στιγμή του συμβουλίου. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι η Σύνοδος Κορυφής της Ρήγας θα είναι επιτυχής. Είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες και των ε, έξι χωρών θέλουν ευρωπαϊκές προοπτικές ή βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κάτι πάρα πολύ θετικό. Θυμάμαι πώς ήταν η κατάσταση για μας εδώ και μερικές δεκαετίες όταν ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γι' αυτό θέλω αυτή η Σύνοδος Κορυφής να είναι επιτυχής και πιστεύω πραγματικά ότι οι προτεραιότητές μας θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ειρήνης και να υπάρχει οικονομική συνεργασία με τις χώρες της ανατολικής ε, γειτονίας αλλά και οι όροι που καθορίζουμε θα πρέπει καταρχάς να είναι οι ευρωπαϊκές αξίες και μετά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και των συστατικών στοιχείων της κοινωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εχθρούς, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα εναντίον της Ρωσίας. Αντιθέτως μάλιστα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ε, συνεργασία, θέλουμε όλοι να είναι εταίροι μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λουκάσοβιτς έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, καταρχάς, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι σήμερα στη συγκεκριμένη αυτή συζήτηση εκφράζομαι εκ μέρους της ύπα της εκπροσώπου Αντιπροέδρου κυρίας Μογκερίνη λάβετε το υπόψη σας παρακαλώ ταυτοχρόνως ως εκπρόσωπος της Προεδρίας υπογραμμίζω ότι αρκετοί επίτροποι ήδη σήμερα βρίσκονται στη Ρήγα, διότι υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις. Η πρώτη διάσκεψη των μέσων ενημέρωση για την Ανατολική Γειτονία κάτι έχει ήδη ξεκινήσει. Σαν Προεδρία εκτιμούμε την άριστη συνεργασία που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής και είναι πολύ σημαντικό που ήδη παρίστανται πολλοί επίτροποι στη Ρήγα. Επανερχόμενοι τώρα στη συζήτηση, επιτρέψτε μου εκ νέου, εκ μέρους της είπα της εκπρόσωπου, να υπογραμμίσω ότι ακούσαμε προσεκτικά όλα τα υποθέντα σήμερα. Ακούσαμε τη συζήτηση και στε βέβαιοι ότι θα λάβουμε υπόψη όλα τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας. Ας επαναλάβω ότι η σύνος Κορυφής της Ρήγας θα αποδείξει ότι η εταιρική ανατολική σχέση παραμένει ε, στόχος μας. Θέλουμε να στείλουμε τα σωστά πολιτικά μηνύματα ότι καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη να προχωρήσει στην εταιρική αυτή σχέση και θέλει να επιδιώξει στενότερες σχέσεις με ανεξάρτητα και κυρίαρχα κράτη που είναι εταίροι της με τι ιδιαιτερότητε του κάθε κράτου να λαμβάνονται υπόψη. Θα δίνουμε υποστήριξη στου εταίρου εκείνου που έχουν αναλάβει τον εκδημοκρατισμό και κάνουν φιλόδοξε ε, αλλαγέ ε, σύμφωνα με τι συμφωνίε ε, σύνδεση. Σημειώνει αυτή η σύνδεση κορυφή ένα νέο επίπεδο των σχέσεών μα με του εταίρου μα. Έχουμε τώρα τις διμερείς μας σχέσεις ε, σύνδεσης, τις διμερείς μας συμφωνίες σύνδεσης με τους εταίρους. Η εταιρική σχέση αφορά έξι χώρες εταίρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ολιστική η προσέγγιση μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να είναι σε επαφή με όλους εταίρους. Ανεξάρτητα με το επίπεδο της σχέσης της κάθε χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, θα αυξήσουμε τις στατικές μας προσπάθειες επικοινωνίας για να εξηγήσουμε ποιε είναι οι σχέσει με τους εταίρου. Περί τίνος πρόκειται. Και τι δεν αφορά αυτή η εταιρική σχέση. Και θα επιχειρηματολογήσουμε λέγοντας ότι δεν απευθυνόμεθα κατά κανενός τρίτου μέρους. Θα συνεχίσουμε συνεπώς το διάλογο με εκείνους που αμφισβητούν τη θέση μας αυτή. Αρκετοί από εσά θέσατε και ένα άλλο θέμα. Ποια είναι η ευρωπαϊκή προοπτική για τη Γεωργία, για τη Μολδαβία, για την Ουκρανία. Και πώς λαμβάνονται υπόψη αυτές οι πτυχές στη διακήρυξη της Ρήγας. Να τονίσω καταρχάς ότι αυτή η κοινή διακήρυξη τη Συνόδου Κορυφή τη εταιρική αυτή ανατολική σχέση είναι κάτι που συνεχίζεται. Εξετάζουμε τη διατύπωση. Συμμετέχουν όλοι. Και τα κράτη-μέλη μα και οι εταίροι μα στη διαμόρφωση του κειμένου. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Γι' αυτό θα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα αυτών. Θα πρέπει η συνένεση να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας, τις προτεραιότητες κάθε χώρας, τις προσδοκίες της και τα κοινά ε, συμφέροντα που έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως βέβαια. Χρειάζεται πραγματιστική αξιολόγηση των προσεπίτευξης στόχων τα επόμενα έτη. Σε αυτό το πλαίσιο η Ρήγα θα πρέπει να τονίσει πρωτίστως ότι πρέπει να κινηθούμε και μπορούμε να κινηθούμε σε νέο επίπεδο σχέσεων με τους τρεις εταίρους μας. Με αυτούς υπογράψαμε τις πλέον φιλόδοξες διμερείς συμφωνίες σύνδεσης. Δείχνει και ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για συμφωνίες με άλλες χώρες που θα ταιριάζουν συμφωνίες με τις άλλες χώρες, με τυτερότητες και θέλουμε να έχουμε ένα γενικό σφαιρικό πλαίσιο που θα χωρά όλους. Πιστεύω λοιπόν ότι κοινή πεποίθηση είναι ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφής. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο χρόνο προς συζήτηση διαφόρων θεμάτων λεπτομερέστερα. Όμως, σεβόμενοι το πρόγραμμά σας, θα φυστώ του χρόνου και κλείνοντας, θα τονίσω ότι εκτιμώ τα μάλα την δέσμευσή σας να στηρίξετε την εταιρική σχέση, την ανατολική. Οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και ο ρόλος αυτών για να παγιωθεί η εταιρική αυτή σχέση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί πρέπει να βοηθήσουμε τους εταίρους να υλοποιήσουν τα όσα μπορούν, τα όσα είναι στις δυνατότητές τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας για την πολιτική, για την ανατολική γειτονία και ευχαριστώ πολύ που νοιάζεστε. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι επιτυχής η Σύνοδος Κορυφής στη Ρήγα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σε ευχαριστώ κυρία μου.